έκθεση Κάμπριλ για μια νέα ΚΑΠ διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολιτών σχεδίων. Το λόγο λοιπόν έχει ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις εισφορές των συναδέλφων, να ευχαριστήσω επίσης τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για την επιτυχία αυτής της έκθεσης τα τεχνικά μέτρα και τα πολιτικά σχέδια είναι τα βασικά εργαλεία για να πετύχουμε τους στόχους της κοινή αλληλευτικής ε, πολιτικής και δεν θα πρέπει να μας ε, ε, παραπλανεί η έννοια των τεχνικών μέτρων ως δευτερογενούς έννοιες. Πρόκειται για μια έννοια με σημαντική πολιτική αξία διότι πραγματικά καθορίζουν το βίο πολλών χιλιάδων αλλιέων. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ε, και να ε, χαραχθεί μια νέα κοινή ελευτική πολιτική, η οποία να συμπεριλαμβάνει μια πρόληψη για τις απορρίψεις. Αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει μια πλούστευση ε, των κανόνων που είναι πλέον παροχημένοι καθώς και εκείνων των κανόνων που είναι λειτουργική και βεβαίως θα πρέπει να εξυπηρετήσει για να βελτιώσει την ε, κατανόηση όλων των νομοθετικών ε, κειμένων τα οποία βρίσκονται σε ισχύ αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση. Ο νέος κανονισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με ευελιξία στις ε, αλλαγές και να λάβει υπόψη την εξέλιξη πιο ε, ευέλικτων ε, μεθόδων ε, αλίας. Και θα πρέπει να βασίζεται βεβαίως σε εγκεκριμένε επιστημονικές βάσεις ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος δυναμισμός όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων και την συμμετοχή των ίδιων των αλλίων στην λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ορθολογική διαχείριση της αλίας. Ε, θα πρέπει να έχουμε ένα ευέλικτο πλαίσιο το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των περιστάσεων και στις νέες ε, προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε ανα πάσα στιγμή. Και θέλω να σα επιστήσω την προσοχή στη σημασία ε, που έχουν τα κριτήρια της αναλογικότητας για να αποφύγουμε δυσμενείς, κοινωνικο... δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις. Η έκθεση αυτή προτείνει μια νέα αρχιτεκτονική του κανονισμού σε τέσσερις άξονες. Τρεις εξ αυτών αφορούν ένα σύνολο κοινών ε, κανόνων, ε, ειδικού ε, κανόνας για τα συνολικά επιτρεπόμενα λεύματα και για τα και ένα τέταρτος άξονας αφορά τα περιφερειακά μέτρα τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές. Ε, οι ετήσιε ποσοστώσει είναι το πιο κατάλληλο όχημα για να γίνονται ε, διαφοροποιήσει σε διάφορα είδη αλίας. Είναι αναγκαίο οι συνομοθέτες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τα πολιετή σχέδια σε σχέση με τις θεσμικέ αλευτικές ικανότητες που προβλέπονται από τη συνθήκη και στη βάση της ε, θαλάσσιας νομολογίας. Θα πρέπει επίσης να αυξηθεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά την εξέλιξη αυτών των προγραμμάτων και σε περιφερειακό πλαίσιο. Και ελπίζω η έκθεση αυτή να συμμετάσχει σε μια επικοδομητική συζήτηση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε όλους τους ε, ενδιαφερόμενους ε, τομείς και να μεριμνήσουμε για την διατήρηση των αποθεμάτων. Ε, ελπίζουμε η πρόταση της Επιτροπής ε, να λάβει υπόψη της ε, αυτές τις βασικές αρχές και τις συστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στη διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Θα σας δώσω όλον τον λόγο γιατί είστε λίγοι και έχουμε και χρόνο. Ο κύριος Μιλαν είναι ο πρώτος ομιλητής. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Μιλαν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια κύριε Μάτο για την έκθεσή σας. Ε, η τροποποίηση του κανονισμού των τεχνικών μέτρων είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις πολύ σημαντικές καινοτομίες που εισήγαγε η νέα κοινή αλληλευτική πολιτική. Παραδείγματος χάρη την απαγόρευση των απορρίψεων. Επίση, ένα νέο κανονισμό των τεχνικών μέτρων θα δώσει ένα τέλο σε αυτή τη διάχυση που έχουμε στην νομοθεσία αυτή τη στιγμή και έχουμε πάνω από 30 κανονισμού του οποίου είναι κατανεμημένα τα μέτρα. Πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο για κοινού κανόνε ε, για όλε τι διαδικασίε και μέσω τη διαδικασία συναπόφαση και μέσω τη περιφερειοποίηση να καθορίσουμε ποιοι κανόνε θα πρέπει να είναι περιφερειακοί και θα μπορούν να αλλάζουν πιο συχνά ώστε να έχουμε και μια κάποια ευελιξία. Όπω είπε και ο κύριο Μάτο, ο τομέα θα πρέπει επίσης να συμμετέχει και στη διαδικασία της ε, ε, ε, τροποποίησης. Επίσης, οι αλλαγές θα πρέπει να βασίζονται σε αυστηρές μελέτες που θα λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές συνέχειες αλλά και την οικονομική και κοινωνική διάσταση της αλίας. Πρέπει να αποφύγουμε σφάλματα του παρελθόντος όπως για παράδειγμα την προηγούμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πλήρη απαγόρευση των παρασυρώμενων δικτύων. Ολοκληρώνοντας να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Μάτε. Ο κύριος Σεράος Άντος. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι η ευρωπαϊκή ελευθερική πολιτική θα πρέπει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις στον τομέα της αλίας και θα πρέπει ασφαλώς να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για την ελευθερική ε, πολιτική του επόμενου, του επόμενου έτους. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειε που είναι σοβαρέ και για το βραχυπρόθεσμο πλαίσιο. Ενδεχομένω δεν υπάρχουν και ε, ανεπανόρθωτες ε, ζημιές σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο για τους αλληλείς. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα σύμφωνα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον ε, εισηγητή τον κύριο Μάτο για τη συνεργασία του. Θα πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ με όλες τις λεπτομέρειες, αλλά συμφωνούμε απόλυτα με την, ε, τον απότερο σκοπό. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν για την βιωσιμότητα και της ελευθερικής πολιτικής και της, ε, του θαλάσσιου περιβαλλοντός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα πρέπει λοιπόν τα τεχνικά μέσα να προσαρμοστούν στην, στις ιδιαιτερότητες κάθε αλληλευτικής περιοχής. Αυτό θα μας οδηγήσει σε μια βιώσιμη αλία. Ο στόχος λοιπόν είναι κοινό, αλλά δεν μπορούν οι λύσεις να είναι καθολικές. Και είμαι... Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεται αυτό ο εισήγητης. Υπάρχουν ακόμα περιοχές στην Ευρώπη όπου η αλία δεν είναι μόνο μια μεγάλη ένας μεγάλος οικονομικός κλάδος, αλλά ένας τρόπος ζωής, ε, μια παράδοση η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί. Οι κανόνες λοιπόν που περιλαμβάνονται για την βιωσιμότητα του αλληλευτικού περιβάλλοντος και του θαλάσσιου περιβάλλοντος που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα μέσων θεωρούμε ότι έχουν, σημαντικά, έχουν λάψει σημαντικά τις ε, παραδόσεις και τον τρόπο ζωής και στην Κροατία. Αυτό δεν θα πρέπει λοιπόν να το επιτρέψουμε. Θα υποστηρίξω το ψήφισμα αυτό γιατί θεωρώ ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι ευγνώμων προς, την, τον Γκάμπριελ Μάτο, ο οποίος ε, έφερε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο, ούτως ώστε εμείς να μπορούμε ε, να, ε, να ξεκαθαρίσουμε τη δική μας θέση πριν ε, υποβάλει η Επιτροπή τις δικές της προτάσεις. Και υπάρχει μία απόσταση μεταξύ της αλίας μικρής κλίμακας και της αλίας που ανοιχτής θάλασσας. Όταν υπάρχει μία πνής, να σημειώνει επακριβώς ε, ε, ε, ποιες, είναι ακριβώς οι ημέρες αλίευσης. Υπάρχουν ορισμένα δίχτυα τα οποία δεν λειτουργούν στην μικρή κλίμακα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε απολύτως ξεκάθαρους ορισμούς. Ούτως ώστε να υπάρχουν τους ποσοστώσεις, την ε, περιοχή αλίας, ε, το μέγεθος των ε, ματιών και επίσης ένα ελεγκτικό όργανο το οποίο να ελέγχει τα αλλιεύματα και τον, την εκφόρτωσή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Στην κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ομοιογένεια, καθώς τα τεχνικά μέτρα βρίσκονται διάσπαρτα σε 30 και πλέον ειδικού κανονισμούς, συνιστώντας ένα περίπλοκο, ετερογενές και ανοργάνωτο σύστημα διατάξεων οι οποίε όχι μόνο δεν διαθέτουν συνοχή αλλά είναι επίση πολλέ φορέ και αντιφατικέ μεταξύ του. η γεωγραφική προσέγγιση των τεχνικών μέτρων αποτυπώνει με σαφήνεια τη διαφορετική μεταχείριση τη μεσογείου καθώ η επιτροπή στην πρόσφατη μελέτη τη για τεχνικά μέτρα δεν συμπεριέλαβε τη μεσόγειο λόγω τη πολυπλοκότητάς τη. έτσι για μια ακόμη φορά βλέπουμε την ευρώπη των δύο ταχυτήτων την ευρώπη του πλούσιου βορρά και την ευρώπη του φτωχοποιημένου νότου θα πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή ένωση να μην διαχωρίζει την κοινή αλληλευτική πολιτική της και να θεσπίζει ισότιμα μέτρα για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υποστηρίξει οικονομικά του φτωχοποιημένου αλληλείς τη Πατρίδα μου τη Ελλάδο, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά λόγω του δυσβάστακτου τρίτου μνημονίου που επέβαλε η τρόικα στην ελλάδα καταστρέφοντα τον πρωτογενή τομέα ένα πρωτογενή τομέα στον οποίο οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στην φόρομπηχτική πολιτική τη Τροϊκα και τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλ. ευχαριστώ. Ο κύριο Κέλλη, ευχαριστώ. Με ενδιαφέρει το θέμα αυτό γιατί ε, κατάγομαι από την Ιρλανδία. Έχουμε πολλά νησιά και πολλούς ανθρώπους ε, σε παράκτιες περιοχές οι οποίοι εξαρτώνται από την αλληλεία για την επιβίωσή τους. Αλλιεύουν εδώ και αιώνες και δυστυχώς ε, έχουν πληγεί λόγω των ευρωπαϊκών πολιτικών ή τουλάχιστον έτσι μου λένε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να τίνουμε ευήκονους αυτά που έχουν να μας πούνε. Όταν τροποποιούμε την ευρωπαϊκή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να ακούμε και την άποψη των ίδιων των αλλιέων, κυρίως αυτών οι οποίοι αλεύουν με μικρά ιδιόκτητα σκάφη. Νομίζω ότι έχουν την εντύπωση ότι κανείς δεν τους ακούει, ιδίως ε, όταν εξετάζουμε θέματα ε, προόδου πρέπει να μπορέσουμε να τους δώσουμε περισσότερες δυνατότητες να αλλιεύουν και ταυτόχρονα να είμαστε δίκαιοι απέναντί τους διότι εξαρτώνται από αυτόν τον τρόπο ζωής και η όλη κοινότητα εξαρτάται από αυτόν τον τρόπο ζωής. Ο κύριος ε, Περέιρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα τεχνικά μέτρα και τα πολιετή σχέδια είναι χρήσιμα εργαλεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλες ε, δυνατότητες ε, στην αλία. Τα πολιετή σχέδια επιτρέπουν μια κάποια σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε ένα τομέα ο οποίος έχει πληγεί όπως ελάχιστοι τομείς με μεγάλη, από μεγάλη αστάθεια. Πρέπει όμως ε, να γίνεται και μια διαχείριση των σχεδίων αυτών με βάση τον τομέα όπου τα κράτη-μέλη θα έχουν και πολύ μεγάλο ρόλο να διαδραματίσουν. Η πρόσφατη αλλαγή της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, που προβλέπει διαχείριση των σχεδίων αυτών ε, μέσω των ε, κεντρικού συστήματος δεν λαμβάνει υπόψη της ε, την ποικιλομορφία που παρουσιάζει ο κλάδος αυτός και όσον αφορά τα αλλιευτικά σκάφη και όσον αφορά τους διάφορους τρόπους αλίας και τους κλάδους αλίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη επικέντρωση στα προγράμματα για να επιτύχουμε τους στόχους ε, να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα αλίας και να ε, καταφέρουμε να επιβιώσουν και οι παράκτιες περιοχές και να διασώσουμε και τα θέματα, Η Επίτροπο. Σας ευχαριστώ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την έκθεση πρωτοβουλίας για τα τεχνικά μέσα ε, διατήρησης του κυρίου Μάτο. Μας δίνει μια πολύ σημαντική ε, παρουσίαση για την απόψη του Κοινοβουλίου για τα τεχνικά μέσα αυτά. Η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ επίκαιρη γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση προετοιμάζει μια νομοθετική πρόταση σε ό,τι αφορά αυτά μέσα για όλη την Ένωση και χαίρομαι ιδιαίτερος που μπορώ να σας πω ότι η έκθεση συνάδει με τη δική μας ανάλυση. Αναγνωρίζει τα θέματα της περιφερειακής διάστασης και της ε, απλοποίησης ως βασικά θέματα. Η νέα λοιπόν αυτή πρόταση είναι προτεραιότητά μας και επιβεβαιώνω ότι σκοπεύουμε να την ε, καταθέσουμε στις αρχές του 2016. Θα περιέχει ένα πλαίσιο βασικών κανόνων που θα καλύπτει όλα τα έντατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτό θα επιτρέψει την περιφερειακή διαμόρφωση και κάποιες ε, αλλαγές οι οποίες ε, σε ό,τι αφορά την ουσία θα αφορούν τη μείωση, μάλλον την μεγαλύτερη ε, περιφερειακή διαμόρφωση. Αυτό θα αποτελέσει λοιπόν την προσέγγιση για την ε, βιώσιμη πολιτική αλληλείας. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δεν θα αλλάξουν τα πρότυπα διατήρησης τα οποία υπάρχουν τώρα και μάλιστα θα βελτιωθούν. Σε ό,τι αφορά τον πολιετή προγραμματισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι συμφωνεί με την ανάλυση της έκθεσης. Αποτελούν άλλωστε ένα βασικό στοιχείο για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής για τους εξή λόγους. Γιατί καταρχάς αποτελούν τα βασικά μέσα για να πετύχουμε τους στόχους της μέγιστης βιωσιμότητας με ένα τακτικό τρόπο. Κατά δεύτερον, συμβάλλουν σε μια σταθερότητα και βεβαιότητα και για τον οικονομικό κλάδο. Και κατά τρίτον, αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την περιφερειακή αυτή διαμόρφωση της πολιτικής. Η διαπραγμάτευση ενός τέτοιου πολιετούς πλαισίου για την Βαλτική προχωρά καλά και καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές θεσμικής φύσεως και πολιτικής φύσεως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει σύντομα να πετύχουμε ένα σχετικό, μια σχετική συμφωνία. Προσβλέπουμε και στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο για τα δύο σημαντικά αυτά ζητήματα που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των γενικότερων στόχων μας περιβαλλοντικής οικονομικής πολιτικής φύσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η σχετική